Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινήσουμε σε ένα λεπτό τη συνεδρίαση και σας παρακαλώ να καθίσετε. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu. Άρχεται η συνεδρία σας κυρίσω την ε, επανέναρξη της ε, περίοδου συνόδου που είχε διακοπεί 11 Νοεμβρίου. Τα κείμενα που έχουν υιοθετηθεί καθώς ε, και τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 11 Νοεμβρίου είναι στη σας. Δεν βλέπω παρατηρήσεις. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις καταρχά. Με μεγάλη ικανοποίηση ενημερωθήκαμε ότι η κυρία Αουν Σανσουτσί έχει απελευθερωθεί. Πρόκειται βεβαίω για την πολύ γνωστή γιατρά τη αντιπολίτευση τη Βυρμανία. Πρόκειται για μία από τι πρώτε πολιτικού, από του πρώτου πολιτικού που τιμήθηκαν με το βραβείο Ζαχάροφ, που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις αγωνιστές της ε, ελευθερίας συνειδήσεως από το 1989. Δυστυχώς δεν έχουμε μπορέσει να την δούμε την ίδια για να τις απονείμουμε, να τις επιδώσουμε το βραβείο αυτό. Εγώ της επέστειλε επιστολή ζητώντας της, εάν έχει την ευκαιρία, να έρθει μέχρι εδώ για να της απονείμουμε το βραβείο σε μια ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 25 Οκτωβρίου έλαβε χώρα, εορτάστηκε μάλλον, η 11η ε, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Οι γυναίκες καθημερινά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, βιασμών, υποφέρουν με διάφορους τρόπους και από διάφορες μορφές καταπίεσης οι γυναίκες. Είναι πολύ υψηλά τα νούμερα των νέων κοριτσιών που θύματα βιασμού κάθε χρόνο και θέλοντας να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτές τις βαρβαρότητες, καταθέτουμε και καταγράφουμε τις, ε, ε, τη βούλησή μας για να περατωθεί κάθε μορφή φυσικής ή ψυχολογικής βίας της βάρος των γυναικών. Άλλε ανακοινώσει. Οι αρμόδιες ισπανικέ αρχές με ενημέρωσαν ότι ο κύριος Ραμόν Χαουρεγκούι Ατόντο αντικαθίσταται από την κυρία Μαρία Ιριγκόιεν Πέρε από 16 Νοεμβρίου του 2010. Καλώς ορίζω τη νέα συνάδελφο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι. Υπενθυμίζω δε ότι δυνάμει το άρθρο 3 παραγραφός 2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο δεν έχουν επαληθευθεί ε, οι συνθήκες εκλογής ή όσο δεν έχει γίνει επαλήθευση ενδεχόμενης ένστασης, η κυρία Μαρία Ιριγκόιεν Πέρες, ε, εδρεύει μέσα στο κοινοβούλιο και στα λοιπά του όργανα, έχοντας πλήρη δυνατότητα άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι έχει εντωμεταξύ καταθέσει τη δήλωση πως δεν ασκεί δραστηριότητα ασύμβατη με το λειτουργήμα του Ευρωβουλευτή. Επίση, θέλω να σα ενημερώσω ότι ο κύριος Κλάουδιο Σύπριαν προσχώρησε στην ομάδα τη προοδευτική συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 15 Νοεμβρίου του 2010. Σα ενημερώνω επίση πω ο κύριος Σπίνο Αρλάκη προσχώρησε στην ομάδα τη προοδευτική συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 18 Νοεμβρίου του 2010. υπογραφή πράξεων που υιοθετούνται υπό τη συνήθι νομοθετική διαδικασία. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με τον πρόεδρο του Συμβουλίου πρόκειται να ε, συνυπογράψουμε 14 ε, πράξεις νομοθετικές που υιοθετήθηκαν υπό τη συνήθι νομοθετική διαδικασία ε, δυνάμει του άρθρου 74 του κανονισμού του Κοινοβουλίου και θα δημοσιευθούν οι πράξεις αυτές στα πρακτικά της περίοδου συνόδου ε, τη παρούσα περίοδου συνόδου είναι στη διάθεσή σα για ενημέρωση και πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή. Τώρα προχωρώ στι τροποποιήσει τη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου, δυνάμει του άρθρο 137 του κανονισμού. Για τη Δευτέρα, γιατί θα κοιτάξουμε κάθε μέρα με τη σειρά από την η διάταξη. Στη Δευτέρα λοιπόν οι πολιτικές ομάδες προτείνουν η συζήτηση για την έκθεση του κύριου Μπερλενγκουέρ ως προς τις ε, πτυχές του προγράμματος δράσεως εφαρμογή του προγράμματος Στοκχόλμη επί του αστικού εμπορικού οικογενειακού και ιδιωτικού, και δικαίου ε, να φύγει από την ημερήσια διάταξη, να μην ε, συζητηθεί στην ημερήσια διάταξη και θα, να ψηφιστεί απευθείας αύριο. Θα εξεταστεί λοιπόν η έκθεση αυτή, αλλά χωρίς συζήτηση, μόνο με ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω. Μας ενημέρωσαν όλες οι πολιτικές ε, ομάδες ότι την πρόταση αυτή, η έκθεση Berlinguer, να μην ε, συζητηθεί και να περάσει τη στην ψηφοφορία, τις ε, βρίσκει όλες σύμφωνες. Για την τρίτη δεν έχουμε καμία τροποποίηση. Κύριε Σούλτς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, για την τρίτη η μερίσια διάταξη αναφέρεται σε έξι εκθέσεις του κυρίου Ματέρα, της κυρίας διορθώνει ο μιλητής, για τη χρήση του ε, Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για την ε, αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης